Well, colleagues, we Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Και μια και έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και κινδυνεύουμε να μην προλάβουμε να εξετάσουμε τις, να ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για όλες τις εκθέσεις όπως έχουν ζητηθεί. Σας προειδοποιώ ότι αν δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε σε μισή ώρα Κάποιες από τις επεξηγήσεις ψήφου θα αναβληθούν για μετά την αυριανή ψηφοφορία. Παντώ σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη γραπτή επεξήγηση ψήφου. Είτε λοιπόν ε, δεν προλαβαίνετε τώρα, είτε προτιμάτε να πάτε να φάτε, αντί να καθίσετε να κάνετε προφορική επεξήγηση ψήφου, να θυμάστε ότι μπορείτε να μας αποστείλετε γραπτή επεξήγηση. Ξεκινώ με την έκθεση Μπαλτσάνη. και τον προπολογισμό 2012, διαφορετικό προπολογισμό. Η κυρία Ανδρίκη Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πριν από ένα χρόνο υιοθετήθηκε ο προπολογισμό του 2012, αλλά ήδη δηλαδή τότε γνωρίζαμε ότι θα ήταν ελληματικό. Και φέτο, στο τέλο του χρόνου, έμεινε σε μόνη επιλογή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ε, πρόταση ενός ορθωτικού προϋπολογισμού για να καλύψει τα 9 δισεκατομμύρια που λείπουν για την κάλυψη των ανηλυμένων υποχρεώσεων. Όμως μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν από τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι τα υπόλοιπα 3 δις θα συμπληρωθούν στις αρχές του προσεχούς έτους καθήκον κοινό και πρόκληση για τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Η εμπειρία όμως από τον προϋπολογισμό του 2012 δίνει πολύ ε, δυσάρεστα και ανησυχητικά μηνύματα. Υπάρχουν, ξέρουμε, εξηγήσει, δικαιολογίε μάλλον, οικονομική κρίση και το καθεξής. Αλλά εάν ο κόσμος χάσει την εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη, τότε η κρίση θα επιδεινωθεί. Ο κύριος Ντανιέλ Χάναν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν ε, ο, ο όταν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έβγαλε το μεγάλο του στινόπρο από λίγη ώρα και υπέγραψε μεγαλοπρεπός τον προπολογισμό του 2013, κατέστημεν όλοι μάρτυρες ενός ε, πολύ εντυπωσιακού ε, επεισοδίου δραματικής τέχνης. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ως προς τις δημοσιονομικές προοπτικές, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, ενώ ο προπολογισμό κάθε χρόνο, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό αυξάνεται μέρα με τη μέρα είναι σαν το σύστημα του ποδηλάτου, ότι πρέπει να συνεχίσει να κάνει πετάλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά θα πέσει. Βέβαια, εγώ θα έβλεπα μάλλον παραλληλισμό με τον κολυμβητή που κυνηγάει ένα καρχαρία και πρέπει να συνεχίσει να κολυμπάει για να μην πέσει βορρά στι ωρέξει του καρχαρία. Εν πάση περιπτώσει όμω, έχουμε διάφορου εδώ καρχαρίες ε, όπως ε, εργολάβους, υπεργολάβους και άλλους που έχουν φτιάξει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα και μάλλον θα τα αφήσουν να καταρρεύσει. Ευχαριστώ. κυρία Μπασέσκου. Πρόεδρε, η ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να εξασφαλιστεί, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει που έχουν αναλυφθεί για το 2012 και να πληρωθούν τα οφειλόμενα ποσά. Γι' αυτό υπερψήφισα αυτή την πρόταση. Η πολιτική συνοχή και άλλα σημαντικά προγράμματα της Ένωσης όπως το Εράσμος κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς κονδύλια στους τελευταίους ε, μήνες του χρόνου. Γι' αυτό χρειάστηκε να κατατεθεί ο διορθωτικός προπολογισμό. Οι μειώσει των δαπανών της Ένωση πιστεύω ότι θα πρέπει να επηρεάζουν τις πιο ουσιαστικές πολιτικές της Ένωσης και όταν έχουμε πολύ ψηλή ανεργία των νέων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να έχει επαρκή πρικοδότηση. πρικοδότηση. Αντίστοιχα, χρειάζεται να υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις υποχρεώσεων, άλυψης υποχρεώσεων αλλά και πληρωμών για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για το προσοχή έτος. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Λαβία και του κυρίου Βόν για το Γενικό προπολογισμό της ευρωπαϊκή Ένωσης και το Οικονομικό του 2013. κυρία Γκέρλινγκ έχετε στο λόγο. Όχι, δεν την θέλετε. Καλώς. Θα ακούσουμε τον επόμενο μιλητή, ο κύριος Ιακολίνου. Είστε εδώ. Ωραία λοιπόν, επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ τη έκθεση για, το νέο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό το 2013, γιατί θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο έκανε επίδειξη αίσθηση ευθύνη σε αφιολογία σε ότι αφορά μια συνέχεια η οποία δεν μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία. Σε ό,τι αφορά την αρχική ανάγνωση υπήρξαν ορισμένα ανοίγματα. Παρά όλα αυτά η συμβολή της Επιτροπής δεν βρίσκεται απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες μας. Η συμφωνία για το πακέτο εγγυάται ορισμένες πολιτικές προτεραιότητες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και που, βρίσκ, και που συνάδουν με τη στρατηγική 2020. Από το, ως εισηγητής θεωρώ ότι επί των εσωτερικών υποθέσεων έχουν γίνει πάρα πολλές περικοπές. Παρ' όλα αυτά η ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκής πόρους για να υπάρξει εγγύηση για τα νέα προγράμματα έρευνα και υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κατάρτιση είναι εκείνο που πριτανεύει. Ευχαριστώ. Κύριο Γιάρη είναι εδώ. Ωραία. Αν δεν είναι εδώ μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Αντρίκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίναμε ένα νέο προϋπολογισμό για το 2013 και πάλι ένας προϋπολογισμός ελλημάτων γιατί οι υποχρεώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υψηλότερες από ε, τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του 2013 είναι πιο περιορισμένος από του 2012. 9% του χαμηλότερου του ΕΠ. Ο προϋπολογισμός σε ό,τι αφορά τις πληρωμές είναι 0,6% υψηλότερο σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν μπορεί να μας ευχαριστεί το γεγονός ότι οι πιστώσεις είναι υψηλότερες το 2013 από ότι το 2012 η αύξηση της ανταγωνιστικότητας χρηματοδοτηθεί καλύτερα με 4,8% αύξηση ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα τύχει χρηματοδότηση με το δότης κατά 6,4% σε σχέση με το 12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι θα μας λείψουν τα κονδύλια του προπολισμού. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συνεπώς, θα πρέπει να εποπτεύσουμε και να θεωρήσουμε τον προϋπολογισμό. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Κυπριακή Προεδρία που μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτό το περίπλοκο πλέγμα ζητημάτων το σχετικό με τον προπολογισμό του 2013. Ωστόσο, ο προπολογισμό αυτό στηρίζεται σε δεδομένα του 1950 σχετικά με την ασφάλεια στην προμήθεια τροφίμων και τι ε, επιδοτήσει στην γεωργία. Όλα αυτά είναι παροχημένα, όπω και η έδρα του Στρασβούργου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εάν έκλεινε θα μα ε, ξεκονομούσε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην κάθε πενταετία. Ενώ συνεχίζονται λοιπόν οι πολιτικές, θα πρέπει να συνεχίζονται οι πολιτικέ και ενίσχυση μόνο για τι πιο φτωχέ χώρε, θα πρέπει τα κονδύλια να αφιερωθούν στι νέε τεχνολογίε, στην ανάπτυξη, την τη ε, τηλεπικοινωνία και γενικότερα τι υποδομέ. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση τη κοινή γεωργική πολιτική, που έχει πολύ μεγάλο προστό του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ε, και να προσαρμοστούν βέβαια και οι μισθοί σε σχέση με αυτά τα οποία ξέρουμε ότι παίρνουν οι ευρωκράτες με τους παχυλούς μισθούς. Όλα αυτά θα έπρεπε να ενσωματωθούν στον προπολογισμό του 2013. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο έχει το λόγο. Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσει του προπολογισμού αυτό έχουν αρχίσει να μετατρέπονται σε φαρσοκομωδία, ενώ χρειάζονται κάποια δισεκατομμύρια ευρώ και δεν τα καταβάλουν οι τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καταβάλει τα ποσά που οφείλει, ενώ πιέζεται και με τον προϋπολογισμό του 2013. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο αυτό τις προκλήσεις της κρίσης, την ανεργία δηλαδή, τα προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα και χρειάζεται φρέσκο χρήμα για να καλύψουμε τις ανάγκες για τα τέλη του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρητά προσπάθησε να διασώσει αυτόν τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάναν. Πρόεδρε, Κάποιο ε, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι το ευρώ που δαπανάτε στι Βρυξέλλε αξίζει πιο πολλά από ότι το ευρώ που θα δαπανηθεί στην κάθε χώρα μέλο. Έτσι φαίνεται να πιστεύουν ορισμένοι. Μα αν είναι έτσι, τότε ε, α του προσλάβουμε όλου ω δημοσίου υπαλλήλου. Α αναλάβει το κράτο το καθήκον ε, και την αρμοδιότητα και την ευθύνη για το κάθε ευρώ που θα δαπανάτε και έτσι λύνεται το πρόβλημα. Μα κοιτάξτε, σα πω, σε εθνικό επίπεδο δεν ε, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με την ε, νοοτροπία αυτή. Γιατί χώρε οι οποίε έχουν τα σοβαρότερα προβλήματα βρίσκονται στη μεγαλύτερη κρίση και με ε, το μεγαλύτερο δημόσιο μηχανισμό ιδιαίτερος. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα δίνουμε περισσότερες εισφορές, περισσότερες συντάξεις, μεγαλύτερους μισθούς, και όλα αυτά για τον κάθε επίτροπο που θέλει να πει στον κόσμο ότι όλα είναι καλά. Μα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλο, μεγάλη αποτυχία, γιατί όσο πιο πολλούς φόρους επιβάλλουμε, τόσο λιγότερη είναι αναδιανομή του δημοσίου χρήματος. Ευχαριστώ κύριε Πασέσκου. Πρόεδρε, η οικονομική κρίση καθιστά κατεπίγουσα την έγκριση του προπολογισμού του 2013. Είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μένα, διότι συμπεριλαμβάνει σημαντικά ε, μέτρα για την ε, εξασφάλιση σύγκληση τη θέση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ο δε νέο προπολογισμό υπογραμμίζει την σημασία του να εκπληρωθούν, να τηρηθούν δεσμεύσει που έχουν ληφθεί στο παρελθόν με τον προηγούμενο προπολογισμό. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ελπίζουμε το έχετε δυνατό. Ο προπολογισμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι δημοσιονομικέ πολιτικέ των κρατών μελών και θα πρέπει να συμπληρώνεται με δράσει με στόχο την, τις επενδύσεις και την οικονομική σταθερότητα. Η δε χρηματοδότηση των πιο σημαντικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωριστεί ω όχι τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε ένα προπολογισμό, ο οποίο κατά αποτελεσματικό τρόπο θα ε, προάγει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κάμπελ. E Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αλλά ξέρετε ότι ο λαός μου ανησυχεί γιατί αυτή τη στιγμή πληρώνουμε καθαρή φορά 30 εκατομμύρια λίρες. Είμαστε στις 118 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, που δαπανώνται μόνο για τη γραφειοκρατία κάθε χρόνο. Και πρέπει να σου πω πως για 18 χρόνια συμβαίνει αυτό στη σειρά. Και τώρα μας ζήτησαν 1,5 δις παραπάνω για φέτος και επίσης για τα επόμενα 7 έτη. Μα με συγχωρείτε, σε ποιο πλανήτη ζούμε στον Πλούτονα, στην Αφροδίτη, στον Άρη, γιατί δεν ζούμε στην πραγματικότητα. Αυτό που είναι ε, πραγματικότητα είναι ο κόσμος στην Ελλάδα υποφέρει, όπου ζει σε συνθήκες χειρότερες από αυτές οι Γερμανίες του 30 λόγω της πολιτικής του ευρώ και των πολιτικών της Ευρώπης. Αυτό ε, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να δαπάνουμε εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να πηγαίνει ερχόμαστε από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες. Πρέπει να κάνουμε περικοπές περικοπές στον προϋπολογισμό και δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω μέχρι να νοικοκυρέψουμε τα δικά μας. Τελειώσαμε την επεξήγηση ψήφου για τον προπολογισμό του 2013 και περνάμε τώρα στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η κυρία Λαρακόνη είναι η πρώτη ε, ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, δεν ψηφίστηκε αυτή η έκθεση και συνεπώς αποσύρω τη δήλωση ψήφου. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη εξήγηση που δώσατε. Η κυρία Ήβα Τζανίκη. Is present? Η κυρία Τζανίκη είναι εδώ. Όχι δεν είναι. Ωραία. Ο λόγος στον κύριο Ζέμκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ψηφίσαμε αυτή την έκθεση και αν κοιτάξετε το σχέδιο της νομοθετικής πράξης θα μπορέσετε να κάνετε μια αναφορά στην Επιτροπή ε, Μεταφορών. Η βασική ιδέα ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εδάφους. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η εγγύηση ε, της ασφάλειας των επιβατών και της πτήσης. Για τον λόγο αυτό κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση ως προς την νομοθετική πράξη. Ευχαριστώ. Με Δυσαρέστησε, με απογοήτευσε κάπω η αντίδραση του συναδέλφου. στόχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στου επιβάτε. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά καθώ και αρκετέ χώρε μέλη και αυτή η προσέγγιση τη ελεύθερη αγορά έχει λειτουργήσει καλά. Τα επίπεδα ποιότητα μπορούν να βελτιωθούν και αυτό εξάλλου προσπάθησα να κάνω. Εμεί πιστεύουμε ότι ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά ε, είναι ο σωστός δρόμος. Η πλήρη άρση των περιορισμών στον τομέα των υπηρεσιών εδάφους θα πρέπει να είναι ο τελικό στόχος. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ε, περιορισμοί. Ε, πιστεύω ότι η αναπομπή μας επιτρέπει να κινηθούμε προς αυτό τον στόχο και να μην, ε, κάνουμε, να μην παλινοδίσουμε σε σχέση με τα όσα επιτεύχθησαν. Κύριο Στάμπλερ. Äh, äh, Πρόεδρε, ε, υπερψήφισα την έκθεση αυτή της Επιτροπής μας με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαφοροποιήθηκα από εκείνους που προτιμούσαν την απόρριψη γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να προφυλαχθούμε από την ε, μανία της απελευθέρωσης. Δεν βελτιώνονται αυτές οι υπηρεσίες εδάφους ε, από την ε, από την απελευθέρωση, από την απορρίθμιση και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Ειδικά στον χώρο των αεροδρομίων είναι πολύ σαφές αυτό. Είναι πολύ λάθος λοιπόν και παράλογο και πολιτικά. Ήδη βλέπουμε ότι οι θέσεις εργασίας στις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια χάνονται λόγω της εισαγωγής εργατικού δυναμικού από αλλού, τότε και η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς πολιτικούς θα είναι πολύ χαμηλή. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνει πιο αποδοτικές αυτές τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης ε, επιβατών και το νομικό πλαίσιο θα ανοίξει περισσότερο την αγορά. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες που θα πρέπει να ξεπεραστούν έτσι ώστε οι επιβάτες να εξυπηρετούνται καλύτερα. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υπηρεσιών και να προωθήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Το άνοιγμα της αγορά αυτών των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει με έναν ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα μεγάλο βαθμό αστάθεια που θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα, θα αύξανε επίσης το κόστος και θα επιβάρυνε ιδιαίτερα τους επιβάτες. Να σε πιστήσω δε την προσοχή στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε ελάχιστους κανόνες, ε, ελάχιστα ε, πρότυπα για τους κανόνες ασφάλειας. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε, λέει ο πρόεδρος, στην επεξήγηση ψήφου για την ε, έκθεση, για την κατανομή των ε, σλότ στα ευρωπαϊκά ε, αεροδρομία. Κυρία Οκόν είναι η πρώτη ομιλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι ότι αυτές οι ρίδες εξασφαλίζουν τη σύνδεση με απομονωμένες περιοχές και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ολοκλήρωσή τους. Η πρόταση εξετάζει θετικά την δημιουργία μιας δευτερογενής αγοράς που ήδη υπάρχει σε ορισμένα αεροδρόμια σε αυτά τα πλαίσια. Κατευθύναμε την παρέμβασή μας προς την ανάγκη να καλύψουμε μια ρυθμισμένη και διαφανή αγορά. Η καινοτομία αφορά τη δυνατότητα μέρος των εσόδων που προέρχονται από την ε, κατανομή των χρονοδιρίδων στην ε, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υπαλλήλους. Βεβαίως υπάρχει ένας κίνδυνος λόγω του ότι οι εταιρείε που έχουν χρονοδυρίες, στα μεγάλα αεροδρόμια τα χρησιμοποιούν για τις ε, πτήσεις μεγάλων διαδρομών και όχι για τις περιφερικές ε, διαδρομές οι οποίες θα αποκοπούν από τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κύριος Μπενιόν, Πρέπει να θυμόμαστε πως η λογική που κρύβει, κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση είναι η προσπάθεια να αποφύγουμε επικαλύψεις ε, και επίσης το γεγονός πως θα διπλασιαστούν οι επιβάτες μέχρι το 2020. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες τέτοιου είδους χρονοθυρίδες ε, μελλοντικά. Θα πρέπει λοιπόν τα μέτρα από αυτά να συνδυαστούν και να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους τρόπους ε, σύνδεσης, για παράδειγμα σιδηροδρομικούς, για να εξυπηρετούνται τα μικρά περιφερειακά κοντινά αεροδρόμια. Επίσης, τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν επιπλέον δυναμικό. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε μεταξύ τους τα διάφορα είδη μεταφορών, να δημιουργήσουμε περισσότερα hub, περισσότερους κόμβους και να κάνουμε περισσότερες πτήσεις μεταξύ κόμβων και όχι σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Θα πρέπει λοιπόν στην εμπορία των χρονοθυρίδων να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε όλα τα όσα είπα προηγουμένως. Η κυρία Μακοβάη έχει ζητήσει το λόγο, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Εάν όχι, μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία Κοστέλο. Ο νέος κανονισμός ε, δίνει και το πλαίσιο για την δευτερινή εμπορία αυτών των χρονοθυρίδων. Και θα ήθελα να σας πω τι συμβαίνει στην Ιρλανδία. Η Air Lingus έχει 23 σλότ στο Χήθρο και επειδή είναι μεγάλη συμφόρηση σε αυτό το αεροδρόμιο, η αξία αυτών των σλότ θα αυξηθεί πολύ στο μέλλον. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ε, τι γίνεται με την πρώτη εξαγορά της Air Lingus από την Ryanair. Νομίζω πως ο κανονισμός αυτός θα παροτρύνει την ε, Ryanair ε, αν αποκτήσει την Air Lingus να πουλήσει τα σλότ στο χωρίς να λαμβάνει υπόψη στρατηγικές ανάγκες της Ιρλανδίας. Ε, και αυτό είναι οι συνδέσεις μεταξύ Δουβλίνου και Χήθρου και το γεγονός πως από εκεί περνάνε τα περισσότερα ε, μακρινά μας ταξίδια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει το σημείο αυτό να ληφθεί υπόψη και να δούμε και τα περιφερειακά αεροδρόμια τι θα γίνουν. Η κυρία Πετικά είναι η επόμενη, δεν τη βλέπω, άρα λοιπόν μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μπιέλανο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι για τα... Ε, ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτό αποτελεί μια από τι βασικέ προκλήσει για την πολιτική μεταφορών που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει το θέμα του δυναμικού, υπάρχει το θέμα του ποσοστού πως ε, ε, των αερομεταφορών δεν αυξάνεται το τελευταίο διάστημα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πώ θα έχουμε τι καλύτερε χρονοθυρίδε και τι καλύτερε ώρε άφηξη και αναχώρηση. Τώρα τον ανέβει το κατόφλι για τα σλότ που χρειάζονται για να διατηρηθούν ε, τα ωράρια ή η αλλαγή του αριθμού των σλότ που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είμαστε σίγουροι που μας καλύπτει. Χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, περιορισμοί στην έκθεση, ε, παρόλο που η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει και κάποιες άλλες προτάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλές για τον καταναλωτή. Δηλαδή, ε, τη δευτερηγενή εμπορία νομίζω ότι εκεί μπορεί να έχουμε μια στρέβλωση της κατάστασης και δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσουμε. Επίσης, οι οικονομικές κυρώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες που δεν σέβονται τις χρονοθυρίδες. Εγώ πάντως καταψήφισα ο κύριος Τάνοκ. Ο στόχος αυτής ε, της ε, πρότασης είναι να έχουμε τη βέλτιση κατανομή και χρήση στα αεροδρόμια στα οποία υπάρχουν συμφόρηση και κυρίως στην περιοχή την οποία εκπροσωπώ, το Λονδίνο, που γίνεται τεράστια συζήτηση για την αεροπλοεία και για το πώς μπορούμε να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τα αεροδρόμια μας. Άρα λοιπόν θέλουμε να γίνει καλύτερη κατανομή των σλότ και να γίνει πιο ανταγωνιστική, ε, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές εταιρείε. Αυτό είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν οι αεροπορικές εταιρείε να διατηρούν τα σλότ ΕΟΤ αρκεί να χρησιμοποιούν το 80% της κατανομής αυτών των χρονοθυρίδων κατά την προηγούμενη ακριβώ περίοδο. Όμως αυτό δημιουργεί πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, δηλαδή συλλογή πληροφοριών για την οικονομική αποζημίωση από την πώληση αυτών των χρονοθυρίδων. Επίσης ευαίσθητες εμπεριοκές πληροφορίες, επιπλέον διοικητικά έξοδα για τις αεροπορικές εταιρείε. Και αυτό το κόστος τελικά τελικά θα μεταφερθεί ε, στα εισιτήρια και θα βαρύνει τον καταναλωτή. Γι' αυτό και καταψηφίσαμε. Η κυρία Ντότς είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ω μέλο αυτού του κοινοβουλίου εκπροσωπώντα τη Βόρεια Ιρλανδία, είμαι υπέρ των τροπολογιών σε αυτή την πρόταση, οι οποίε διασφαλίζουν ότι οι αλλαγέ στην κατανομή των χρονοθυρίδων θα αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών και των κεντρικών αεροδρομίων. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η δική μου εκλογική περιφέρεια περιφέρεια θα θυγεί και θα θυγεί και η ευμερία στην περιοχή. Σε μια διαρκώς παγκοσμιοποιημένη αγορά η πρόσβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η προτίμηση ε, στην κατανομή χρονοδυρίδων σε μικρά αεροδρόμια θα ενισχύσει τις επενδύσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για την οικονομία μας. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Μπασέσκου. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής γιατί και εγώ με τη σειρά μου πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στα αεροδρόμια ενώ παράλληλα εγγυάται μια βέλτιστη κατανομή των χρονοθυρίδων. Το σύστημα μέχρι στιγμής απεδείχθη αναποτελεσματικό. Για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα, η εξυγίαση των μηχανισμών και η εφαρμογή τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Παράλληλα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανταγωνιστικότητα των συντελεστών και να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ε, ε, βελτίωσης της διαφάνειας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τις διατάξεις αυτές. Εκτός από αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή την ανεξαρτησία των συντονιστών. Ενώ οι δευτερογενείς αγορές των ε, χρονοθυρίδων θα πρέπει να ρυθμίζεται καλύτερα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λέχτρικ σε ό,τι αφορά την, το προκαλούμενο Θόρυβό τους αερολιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Κόμη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκφράστηκα θετικά για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ε, Συμβουλίου που εισάγει κανονισμού για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάντηση με το προκαλούμενο θόρυβο στους λιμές Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση έχει σκοπό να επικαιροποιήσει τα υπάρχοντα μέτρα και να επιτρέψει στι αρχέ να βελτιώσουν τα πράγματα ω προ το θόρυβο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίζει καθοριστικό ρόλο ε, στον τομέα αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά την ηχητική ρήπαση βρίσκεται πολύ πίσω. Ε, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που θίγονται από το προκαλούμενο θόρυβο και που νιώθουν την υγεία τους να ε, επιδεινώνεται. Τα άτομα που ζουν κοντά στα αεροδρόμια, αεροδρόμια δέχονται μία τριπλή ρήπανση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα των αεροδρομίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζανώνη ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο αυξημένο θόρυβο που έχει σχέση με τι αερομεταφορέ, ιδιαίτερα στι νυχτερινέ πτήσει, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωή 4 ε, εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που ζουν κοντά στα αεροδρόμια. Αυτοί οι πολίτε είναι θύματα μια τριπλή ρήπαση ακουστική, ατμοσφαιρική και χημική. Ο θόρυβο που προκαλείται από τι αερομεταφορέ, κυρίω στι νυχτερινέ, έχει δυσμενεί επιπτώσει στην υγεία. Παράλληλα, αλλά οι περισσότεροι από τους πολίτες που ταξιδεύουν θα επιθυμούσαν να έχουν τη δυνατότητα να, έχουν, επιλέγουν. Δίκως άλλο η παρουσία ενός αεροδρομίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας περιφερειακής ανάπτυξης καθήκων μας είναι να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις και να προβλέψουμε δεχομένους περιορισμούς έτσι ώστε να βρεθεί η σωστή τι ισορροπία μεταξύ των ε, ε, αντικρουόμενων αυτών αναγκών. Όπω υπογράμμισε συχνά η Επιτροπή Περιβάλλοντο του Κοινοβουλίου, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη μόνο του οικονομικού παράγοντε. Η προστασία τη υγεία των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν κοντά στα αεροδρόμια θα πρέπει να είναι ο πρώτιστο σκοπό μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπέν, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για το προκαλούμενο θρόλυβος ε, ε, αερολιμένες. Η προσέγγιση της είναι εξισορροπημένη και λαμβάνονται οι υπόψη οι επιπτώσει του θορύβου στην ποιότητα ζωής αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων ε, υπηρεσιών. Ο τομέα των αερομεταφορών χρειάζεται ασφάλεια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι τοπικέ αρχέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνουμε κάτι παράνομο με βάση το νόμο ε, περί ε, ανταγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε προσεκτικά το, το τμήμα αυτό ψηφίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να δώσουμε στις αεροπορικές εταιρείε μια βεβαιότητα και μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και τώρα κυρία Μακοβέη. Παρακαλώ. Κυρία Μακοβέη. Α, έβλεπα άλλο όνομα στην οθόνη, Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Όπως λέει η Διεθνής ε, Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, τα επηρεαστούν πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων τα επόμενα χρόνια από την χορύπανση που ξύνουν τα αεροπλάνα και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο υποστηρίζω την πρόταση για να περιοριστεί στο, ελάχιστο η ενόχληση των πολιτών τη Ευρώπη που μένουν κοντά στα αεροδρόμια. Πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στι πτυχέ αυτέ. Δεδομένου ότι σε περίοδου κρίση πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ε, ισορροπία κόστου και αποτελεσματικότητα. Πρέπει λοιπόν όλες οι πτυχέ να αξιοποιηθούν. Δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε σφαλμένους υπολογισμούς κόστους και των λοιπόν περιορισμών και γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες και διαδικασίες για απόλυτα ακριβείς αξιολογήσεις της, ε, των μέτρων αυτών, τα οποία θα είναι καταλληλότερα για, για τον περιορισμό της συγχωρήπανης. Ευχαριστώ. Την κυρία Πιετικά είναι να έχω τώρα στον κατάλογό μου, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Και έτσι Δίνω το λόγο στην κυρία Φόρντ. Εγώ, πρόεδρε, καταψήφισα το κανονισμό για του λειτουργικού περιορισμού σε συνάρτηση με το προκαλούμενο θόρυβο ερωτημένο, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσαν πολύ καλύτερα και αποτελεσματικά να είχαν εισαχθεί σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Το να εισάγουμε λοιπόν νομοθεσία μέσω κανονισμού αντί για την οδηγία καθιστά πολύ πιο δύσκολο για το κάθε κράτο μέλο να ε, αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες της κάθε κοινωνίας, θα πρέπει η φωνή τους όταν έχουμε ζητήματα υγείας ε, και δημόσιας υγείας και η χορύπανσης να ε, ακούγεται πάντα η φωνή των πολιτών. Και εγώ υποστηρίζω σε τέτοια θέματα τη διεθνή συνεργασία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την ε, ανάπτυξη και εισαγωγή των πιο καθαρών, πιο πράσινων, λιγότερο ρηπογόνων ή χωριπαντικών αεροπλάνων. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με ένα μέτρο και ένα σταθμό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ ο κύριος Μπιέλλον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα, δρα... αεροδρόμια με τις δραστηριότητε τους προξενούν πολύ, πολύ μεγάλη χορύπανση, θόρυβο που επηρεάζει τις ε, ζώνες γύρω από αυτά και έτσι οι κάτοικοι, οι περίοικοι των αεροδρομίων έχουν πολλά προβλήματα η χορύπανση. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί ένα μηχανισμό αποτελεσματικό για τον περιορισμό τη χορύπανση στι ζώνε γύρω από τα αεροδρόμια. Κάποιε από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ όμω ότι πρέπει αυτέ οι εξουσίε να περιοριστούν μόνο για τι περιοχέ για, τις, ε, για τους τομείς εκείνους που μπορούν να καλυφθούν ε, με κατεξουσιοδότηση πράξης. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να εισαχθεί η ε, δέσμη μέτρων με κανονισμό αντί για οδηγία. Δεν είναι αυτός ο καταλληλότερος τρόπος. Εξάλλου αν κοιτάξουμε τις προϋποθέσεις για την επιλογή του κάθε ενός από τα νομοθετήματα και τα μέτρα που θα πρέπει να εισαχθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν βλέπω γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει με κανονισμό για όλους αυτούς τους λόγους κατεψήφισα. Ευχαριστώ κύριο Σαντονιώτση. Δεν τον βλέπω όμως. Και έτσι... Καλώ την κυρία Ντότς να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως βουλευτής της Βόρειας Ιρλανδίας δεν μπορώ να εγκρίνω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή ε, λειτουργικών περιορισμών στη συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό θα, κατηργού, θα καταργούσε τις διατάξεις της προϋπάρχουσας οδηγίας του 2002 η οποία έχει επιτρέψει στο αεροδρόμιο του Belfast να περιορίσει κατά πολύ ε, αποτελεσματικό τρόπο την χορύπανση που προξενούν τα αεροπλάνα και δεδομένης και της γεωγραφικής του κατάστασης. Είναι ζώντες κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και οι επιχειρήσεις στο Belfast αλλά και στην περιοχή του North Time και γι' αυτό είμαι κατά της πρότασης. Η νέα πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνεται βεβαίως στην νυχτερινή εκπομπή χορύπανσης από τα αεροπλάνα και ιδιαίτερος ζητεί την εισαγωγή λειτουργικών περιορισμών μόνο όπου αυτό χρειάζεται και όπου απαιτείται από την ισορροπία κόστου και αποτελέσματο. Όμω το σχέδιο κανονισμού περιορίζεται στο να εξετάζει μόνο τα αεροδρόμια που έχουν ένα μεγάλο όγκο κυκλοφορία αεροπλάνων και έτσι τα μικρότερα αεροδρόμια δεν αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Ντότ ήταν η τελευταία εγγεγραμμένη στο κατάλογο των επεξηγήσεων ψήφου για την έκθεση του κυρίου Λάιχτφριντ. Τώρα έχουμε ακόμα τρει εκθέσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφοφορία, χωρί όμω να μα μένει άλλο χρόνο για να ακούσουμε επεξηγήσει ψήφου. Και όπω σα είχα πει εξ αρχή, αναβάλουμε ε, τι επεξηγήσεις ψήφου για αύριο μετά τις ψηφοφορίες. Γι' αυτό επιτρέψτε μου τώρα να διακόψω την συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα όπου θα ξαναρχίσει η συνεδρίαση. Και παραλαμβάνω, στην αλφή μπορείτε και γραπτό να καταθέσετε επεξήγηση ψήφου ή προφορικό αύριο μετά τι ψηφοφορίε. Σα ευχαριστώ. Διακόπτουμε έω τι 3 το μεσημέρι.